αστικές κυρώσεις. Το ευρώ είναι σε σαθρά θεμέλια και όχι μόνο αυτή τη βδομάδα, αλλά τελευταία πενταετία Ευρωπαίοι πολιτικοί ε, ασχολούνται με την ελληνική κρίση που δεν είναι ε, κάτι που πλήττει μόνο τους Έλληνες πολίτες αλλά όλους τους πολίτες στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι δημοκρατικό μας καθήκον να εξετάσουμε ε, και να αναδείξουμε όλες τις αιτίες και να βγάλουμε τα διδάγματα και τα συμπεράσματά μας. δεν ε, χρειάζεται ακόμα ένα ψήφισμα, ακόμα μία έκθεση. Χρειάζεται μία σε βάθος ε, έρευνα και να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους. Δεύτερον, πώ μπορούμε να φροντίσουμε οι συμφωνίε για το χρέο και για τον προπολογισμό να τηρούνται επιτέλου. Αν θέλουμε να ενισχύσουμε την ΟΝΕ θα πρέπει να αρχίσουμε από τα θεμέλια, από τη βάση. Δεν έχει νόημα να οικοδομούμε σε σαφρά θεμέλια. Γι' αυτό θα πρέπει επιτέλου οι κανόνε για τον προπολογισμό με διαφάνεια, με αυστηρότητα και με συνέπεια να εφαρμόζονται. Θα πρέπει να δούμε πώς θα εκπονηθεί ένα σύστημα για περισσότερους ε, ανεξάρτητους ελέγχους και αυτόματες κυρώσεις. Πώς μπορούμε λοιπόν να τα ενισχύσουμε όλα αυτά, ειδού η ερώτηση και περιμένουμε μεγάλη περιέργεια να δω τι θα απαντήσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το Συμβούλιο. Ευχαριστώ πολύ. Okay. Ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Μπάλτσα έχει το λόγο για δύο λεπτά παρακαλώ. Με ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Το έτος 2011 ενισχύθηκε το Σύμφωνο Σταθερότητας και Ανάπτυξης. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και η Ευρωπαϊκή επιτροπή από κοινού κατάφεραν τα κράτη-μέλη να μην είναι εκείνα που θα αποφασίζουν από μόνα τους. Τώρα που έχει περισσότερα δικαιώματα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα πρέπει ε, να μπορούμε να υπολογίζουμε σε αυτήν ότι θα τα εφαρμόζει σωστά. Δείχνει η κατάσταση ότι η σωστή τήρηση των κανόνων ε, είναι θέμα επιβίωσης για την ΟΝΕ. Είδαμε ε, η κρίση τι επέφερε και θα πρέπει να βγάλουμε συμπεράσματα. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή φέρει εδώ πολύ μεγάλη ευθύνη. Και σε αυτή την ευθύνη θέλουμε σήμερα ε, ε, να υπενθυμίσουμε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Οι κανόνες για το Σύμφωνο Σταθερότητας και Ανάπτυξης θα πρέπει να ισχύουν εξίσου για όλα τα κράτη-μέλη. Δεν υπάρχουν μεγάλα ούτε μικρά κράτη όταν πρόκειται για χρέος και ελλείμματα. Οι αριθμοί είναι αριθμοί και παραμένουν ακόμα και άμα τους γυρίσουμε ανάποδα. Εμείς δεν δεχόμαστε οικονομικές αναλύσεις να διαστρεβλώνονται ή να ερμηνεύονται κατά το δοκούν. Θέλουμε ε, νυφάλια αντικειμενική αξιολόγηση ε, των κρατών μελών και ανεξάρτητη οικονομική ε, ανάλυση με επικεφαλής αναλυτές που να μπορούμε να διαβάζουμε τις αναλύσεις και με τον ίδιο τρόπο ανεξάρτητα να γίνονται όλα αυτά για όλα τα κράτη-μέλη. Γι' αυτό απευθύνουμε έκκληση στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή να ανταποκριθείτε στο ρόλο σας ως ουδέτερος ελεγκτής του προϋπολογισμού. Πρόκειται για το Σύμφωνο Σταθερότητας και Ανάπτυξης και για τα θεμέλια τα ίδια και τη βιωσιμότητα της ΟΝΕ. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Ευχαριστώ πολύ η Πρόεδρος. Θα ήθελα να παρακαλέσω τους συναδέλφους να κάνουν ησυχία. Θα ψηφίσουμε στις 8 η ώρα. 8 αρχίζουν οι ψηφοφορίες. Γι' αυτό θα πρέπει οπωσδήποτε να συζητήσουμε και ε, αυτό το θέμα της ημερήσιας διάταξης. Ο κύριος Ουρτάσουν. Ε, Ευχαριστώ. Η πολιτική μου θα ήθελε να μάθει ακριβώς ποια είναι τα κριτήρια για την εφαρμογή του Συμφώνου Σταθερότητας και για τα μέτρα της διαφάνειας. Γιατί έχουμε εδώ πολλές πολιτικές ομάδες που θέτουν το ερώτημα γιατί θέλουν μια πιο αυστηρή εφαρμογή του συμφώνου. Το θέμα είναι ότι εδώ έχουμε ε, πάρα πολλές περιπτώσεις κατά τις οποίες αυτοί οι κανόνες αντιβαίνουν στους σκοπούς του συμφώνου. Άρα θα πρέπει να προβληματιστούμε μέχρι ποιο βαθμού αυτή η ευελιξία επαρκεί ή όχι. Γιατί έτσι έχει συμβεί. Χρησιμοποιείται η ευελιξία για να νομιμοποιήσουμε κάποια de facto στήματα, όταν κάποιος δηλαδή κάνει κάποια ζαβολιά, κάποιο κράτος. Επομένως, αυτό θα πρέπει να μας εξηγήσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και αυτό θα πρέπει και να βελτιώσει. Θα πρέπει φυσικά να είναι ξεκάθαροι οι σχετικοί κανόνες, να μας πει η Κομισιόν πώς θα εφαρμοστούν τα κριτήρια ή να μας πει επίση ποια θα είναι η μεθοδολογία πολύ σημαντικό θέμα. Να μας εξηγήσει επίσης η Ευρωπαϊκή Επιτροπή τι είδους οικονομική ανάλυση έχει κάνει, τι έχει κάνει για να δει πώς θα κάνουν να τα τα κρατη Επίσης, τι ανάλυση θα είναι η βάση για τις συστάσεις του Συμβουλίου, ούτω ώστε να τεθεί σε εφαρμογή το six-pack, τα μέτρα τέλος πάντων διακυβέρνησης. Εν κατακλείδη, πότε θα δημοσιεύσετε την νομική γνωμοδότηση του 12 ε, του 15 και έχουμε το ε, επίση τον κασμό του 1049 αυτά είναι πολύ σημαντικά ε, next Κύριο Τζάνι είναι ο επόμενος ομιλητή για δύο λεπτά. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Εγώ θέλω να ξεκινήσω για την ανάλυση μου ε, για κάτι με το οποίο βρίσκει σύμφωνο. Το Δεκέμβριο είπαμε ότι θα πρέπει να λάβουμε υπόψη το τι έκανε ένας καθηγητής και πρώην υπουργό ο κ. Γκαρίνο που ε, επεσήμανε τις αιτίες της κρίσης που συνταράσσει την Ευρώπη και είπαμε το ρόλο του Συμφώνου Σταθερότητος γιατί οδηγήθηκαν τα κράτη-μέλη σε, σε κάποιες παράλογες λύσεις για τα δημοσιομικά τους και επίση δέθηκαν τα κρατημέλη χειροπόδρα με κάποιους κανονισμούς. Οπότε τώρα ε, δεν μπορούμε να πάμε σε, κάποια θετική, ε, σε κάποιο θετικό ισολογισμό. Άρα βλέπουμε ότι δεν βρίσκουμε λύσεις στη σημερινή ε, κρίση. Έχουμε το six pack και το two pack και αυτό το σύμφωνο σταθερότητας. Ε, αυτά φρενάρισαν τις δυνατότητες ανάπτυξης για τα κράτη-μέλη πώς ισοσκελίστηκε ο πληθωρισμός, πώς θα γίνει αυτό η ανάπτυξη. Επομένως βρισκόμαστε σε κάποια ε, αντίθεση με αυτό το οποίο προβλέπουν οι συνήθειες στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Κατεχρόνια το κράτος μέλος δεν προχωράει σε ανάπτυξη. Επομένως να μας πει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πώς ερμηνεύει αυτή την αντίφαση, τι θα κάνει για να άρει αυτή την αντίφαση θα πρέπει να καταφέρουμε να καταλάβουμε το ότι οι κανόνες ερμηνεύονται με κριτήρια πολιτικής βούλησης. Γιατί κλείνουμε τα μάτια στις ζαβολίες Γαλλίας ή Γερμανίας. Ε, είδατε τι γίνεται με το υπερβολικό εμπορικό πλούρασμα της Γερμανίας. Βλέπουμε επομένως το, το ότι τελικά η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι αδύναμη με τους δυνατούς και αποφασιστική και αυστηρή με τους αδύναμους. Φερέιρα. Κυρία Πρόεδρε, κυρία Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι, η ευελιξία που χρησιμοποίησε η Κομισιόν στην εφαρμογή του Συμφώνου Σταθερότητας δεν ε, σημαίνει όπως λένε ορισμένοι ότι έγινε μια κρυφή αλλαγή στους κανόνες οικονομικής διακυβέρνησης. Αντίθετα η ευελιξία αυτή προβλεπόταν από πολύ καιρό από τους κανόνες. Το θέμα είναι ότι η προηγούμενη Επιτροπή για ιδεολογικούς λόγους πιστεύω δεν θέλησε ποτέ να τη χρησιμοποιήσει. Και γι' αυτόν τον λόγο οι Ευρωπαίοι Σοσιαλιστές τώρα υποστηρίζουν την απόφαση της Κομισιόν που επιτρέπει προσαρμογή του Συμφώνου Σταθερότητας σε συγκεκριμένη κατάσταση της κάθε χώρας έτσι ώστε να μην συμβάλλουμε στις καταστροφικές πολιτικές που εφαρμόστηκαν μέχρι τώρα. Και σήμερα επιβεβαιώνουμε ότι χρειάζεται μεγαλύτερη ε, διαφάνεια στην εφαρμογή των κανόνων για να φανεί ποιο είναι το πλαίσιο για τις αναπτυξιακές ρήτρες και τις επενδύσεις. Σε αυτά τα πλαίσια για να υπάρξει λοιπόν μεγαλύτερη διαφάνεια η σοσιαλιστική ομάδα θα ήθελε η Κομισιόν να μας ξεκαθαρίσει μερικά πράγματα. Πρώτον, με ποια μεθοδολογία θα αξιολογήσει τα δημοσιονομικά των κρατών μελών ο, τα πλεονάσματα και την δυνατότητα ανάπτυξης σε ποσοστό του ΑΕΠ. Με τι μέθοδο λοιπόν θα υπολογίσει επαναλαμβάνω και την προστιθέμενη αξία των μεταρρυθμίσεων, των διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων. Και πάλι στο ίδιο θα ήθελα να ξέρω πώς θα υπολογίσει η Κομισιόν τις επιπτώσεις των συστάσεών της στη διαδικασία της σύγκλησης μεταξύ των χωρών μελών. Αν μπορούσε να μου απαντήσει θα της ήμουν ευγνώμων. Κύριε Ματίας, δύο λεπτά. Ευχαριστώ πολύ Πρόεδρε. Όταν κοιτάξουμε το περίφημο SGP βλέπουμε ότι υπήρξε καταστροφικό για την ευημερία των πολιτών μας αλλά επίσης ότι έχει επιβληθεί με τελείως αδιαφανή τρόπο Καμία, κανένας δημοκρατικός χαρακτήρας και διαπιστώσαμε μόνο την αύξηση των χρεών. Ερωτώ λοιπόν την Κομισιόν έμαθαν, πήραν κανένα μάθημα από αυτό ή ακόμη μια φορά θα εφεύρουν ψεύτικα επιχειρήματα για να δικαιολογηθούν. Πότε θα αλλάξει η έμφαση η Κομισιόν για να αναγνωρίσει ότι η λιτότητα έχει αποτύχει πλήρως και ότι χρησιμοποιεί το χρέος σαν πρόσχημα αγνοώντας το γεγονός ότι ακόμα και σε περιπτώσεις που έγιναν μέτρα προσαρμογής Μόνο το ιδιωτικό χρέος ήταν σε εκείνες τις περιπτώσεις το πρόβλημα και όχι το δημόσιο. Είναι διατεθειμένη η Κομισιόν να αρχίσει να τα εποπτεύει όλα αυτά και τα πλεονάσματα. Με σκανδαλίζει, βρίσκω σκανδαλώδη την έλλειψη σοβαρότητας σε αυτούς τους υπολογισμούς της Κομισιόν. Γιατί τελικά απλώς παίρνει τιμωρητικά μέτρα για όσους έχουν υπερβολικά ελλείμματα. Χρησιμοποιεί δύο μέτρα και δύο σταθμά τιμωρώντας τις χώρες που έχουν δυσκολίες. Θα αφαιρέσει επιτέλους τις απαράδεκτες κυρώσεις. Οι χώρες που έχουν υπερβολικά πλεονάσματα και αυτές παραβιάζουν το SGT αλλά δεν έχουν ποτέ τιμωρηθεί. Θέλω λοιπόν να μου πείτε εάν η Κομισιόν είναι διατεθειμένη επιτέλους να σκεφτεί όπως θα έκανε ο κάθε λογικός άνθρωπος ότι οι επενδύσεις δεν είναι το ίδιο πράγμα με τις δαπάνες γενικά και ότι οι χώρες που θέλουν να επενδύσουν δεν πρέπει να εμποδίζονται. Κυρία Σιλβιγούλα, ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Ευχαριστώ κύριε Επίτροπε που είστε παρόν ενώπιόν μας για να ασχοληθούμε με αυτό το λεπτό και ευαίσθητο θέμα της ερμηνείας του Συμφώνου Σταθερότητας και Ανάπτυξης. Είναι δύσκολα, περίπλοκα τα κείμενα. Κύριε Επίτροπε, με ακούτε? Φιλανδικά δεν μπορώ να τα πω, λυπάμαι. Euh, το θέμα λοιπόν ε, που τίθεται εδώ, ευχαριστώ κύριε Επίτροπε, χαίρομαι πάρα πολύ όταν με ακούτε. Είμαι ευτυχής. Ένα από τους λόγους λοιπόν έλεγα που κάναμε αυτή την ερώτηση είναι ότι στην προηγούμενη επιτροπή αγωνιστήκαμε με τον Επίτροπο Όλη Ρεν για να βεβαιωθούμε ότι θα υπάρξει ε, ισότιμη ε, εφαρμογή ε, του Συμφώνου Σταθερότητας και θα ίσχυαν ήδη οι κανόνες προς όλους. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή όταν δέχεται ότι εξαγγέλλονται μεταρρυθμίσεις χωρίς να υλοποιούνται αρχίζουμε να μπαίνουμε σε ένα ολιστηρό έδαφος και δεν γίνεται καθόλου σεβαστή ισότητα μεταξύ των κρατών μελών. Ευχαριστώ. Okay. Thank you. Ωραία, ευχαριστώ. Η κυρία Καλίνα Λούκασεβίτσα, εξ ονόματος του Συμβουλίου, προεδρεύουσα για τρία λεπτά. Ε, κυρία Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, αξιότιμοι κύριοι βουλευτές, να σας ευχαριστήσω διότι με καλέσατε να σας μιλήσω για αυτό το σημαντικό θέμα το θέμα της διαφάνειας σχετικά με την εφαρμογή του Συμφώνου Σταθερότητας το Σύμφωνο Σταθερότητας και Ανάπτυξης είναι πολύ σημαντικό για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης πρόκειται για ένα πλέγμα κανόνων ε, θεσπίζεται έτσι μια σταθερή δημιουργική πολιτική και έτσι έχουμε χρηματοδοτική, χρηματοοικονομική μόλις στην Ευρωπαϊκή Ένωση και όταν ε, αξιολογούμε τους προϋπολογισμούς των κρατών μελών θα πρέπει να δούμε κατά πόσον αρκούν αυτοί οι κανόνες, αν υπάρχει περιθώριο ευελιξίας, αν θα πρέπει να λάβουμε υπόψη τις ιδιοτυπίες, τα ιδιαίτερα χαριστικά της κάθε κράτης μέλας. Ε, για αυτό χρειάζεται κάποιο είδου αξιολογήσεις, ε, στεγανές, και αμερόληπτες. Αυτά τα ζητήματα ε, εθίγησαν και σε παλαιότερες συζητήσεις σε σχέση με την ε, έκθεση Μπερές για την ε, οικονομική διακυβέρνηση. Εγώ τώρα όμως θέλω να σας πω για κάποιες πρόσφατες βελτιώσεις του συντονισμού οικονομικών πολιτικών. Έχουμε μια καινούρια θεσμική αρχιτεκτονική. Αναβαθμίζεται έτσι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Επίσης με τους νέους κανόνες ε, υπάρχει διαφάνεια, υπάρχει υπευθυνότητα ε, από πλευρά των κρατών μελών. Όλα αυτά μπορείτε να βρείτε στην ε, ιστοσελίδα μας. Το Συμβούλιο δε όταν συζητεί βοηθάτε από αναλυτές ανεξάρτητους και αμερόληπτους. Επίσης στηριζόμαστε και σε κάποια έγγραφα εργασίας των υπηρεσιών μας, αλλά στηριζόμαστε και στις πληροφορίες που δίνουν τα κράτη-μέλη. Ιδίως όσον αφορά αυτά τα καινούρια ε, μη υποχρεωτικά μέτρα σε περίπτωση που επιλέγουν να τα υλοποιήσουν τα κράτη-μέλη. Έτσι ζυγίζουμε τις θέσεις των κρατών μελών και προσπαθούμε να καταλήξουμε σε κάποια συμφωνία, σε κάποια ε, συμφωνία λέω, για την δημοσιονομική πολιτική. Αυτό κάνουμε και όποτε έχουμε υπερβολικό έλλειμμα. Αυτό και κάναμε και στην περίπτωση της Γαλλίας. Οι τρεις προτεραιότητες του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου είναι πρώτα απ' να διευκολύνουμε τις επενδύσεις. Δεύτερον, να εφαρμόσουμε διαφορετικές μεταρρυθμίσεις και τρίτον, να μπορέσουμε να καταφέρουμε να υπάρχει υπεύθυνη δημοσιονομική πολιτική. Είναι άλλες λόγες. Πρόκειται για ένα από τα στοιχεία τα οποία επιβάλλεται να μετέλθουμε. Γιατί οι επενδύσεις και οι μεταρρυθμίσεις είναι πολύ σημαντικές. Αυτά τονίζονται και οι Ευρωπαϊκές Επιτροπές. Για το πόση ευελιξία θα πρέπει να έχουμε σε σχέση με ε, το σύμφωνο σταθερότητας. Οπότε θα πρέπει έτσι με ευελιξία να εφαρμόσουμε τις σχετικές διατάξεις. Πάντως, εγκατακλείδη πρέπει να σας πω δύο λόγια για τον ε, γενικότερο ρόλο του Συμφώνου Σταθερότητας και Ανάπτυξης και για το πόσο συμβάλλει στην ολοκλήρωση της ΟΝΕ στις 24 Δεκάτου του 2014 είχαμε μια ευρωπαϊκή συνάντηση κορυφής. Εκεί συζητήθηκαν ποια θα ήταν τα επόμενα βήματα ούτω ώστε να ολοκληρωθεί η Οικονομική Νομισματική Ένωση. Οπότε και φτάσαμε στην έκθεση των πέντε πρόεδρων. Εκεί διατυπώνονται κάποιες συστάσεις βραχυπρόθεσμα, πώς θα ενδυναμωθεί η ΙΟΝΕ, αλλά επίσης προτείνω και κάποιες λύσεις πιο μακροπρόθεσμες. Αύριο το Συμβούλιο πρόκειται να ε, ανταλλάξει απόψεις για αυτήν την έκθεση των πέντε Προέδρων. Προείπα στην σημερινή συζήτηση ότι έχουμε τώρα την προλίανση του εδάφους για το Συμβούλιο και θα πρέπει να κάνουμε ό,τι πρέπει από το χέρι μας για να μπορέσουμε να ε, ε, εξομαλύνουμε την κατάσταση για τις διαφορές των χωρών στην Ευρωζώνη για να δούμε πώς δεν θα έχουμε τέτοιες διαφορές που να ροκανίζουν το μέλλον της Ευρωπαϊκής Ένωσης και είπαμε το πώς θα υλοποιήσουμε τις σχετικές προτάσεις αυτές που διατυπώνουν οι πέντε πρόεδροι στο κείμενό τους. Αγαπητοί κύριε βουλευτές, πιστεύουμε ότι θα μπορέσουμε να συνεχίσουμε να έχουμε κοινό όραμα για το μέλλον της ΟΝΕ και θα μπορέσουμε να υλοποιήσουμε όσο θέλουμε. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρος. Και αξιότιμοι συνάδελφοι, κυρίες και κύριοι, θα σας παρακαλούσα να κάνετε λίγη ησυχία για να μπορέσει να γίνει η συζήτηση. Ναι. και να ακούσουμε τον κύριο Κατάινεν, παρακαλώ. Κυρία Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, η Επιτροπή συμμερίζεται την ανησυχία του Κοινοβουλίου για την διαφάνεια και την εφαρμογή της δημοσιονομικής εποπτείας για περισσότερη ασφάλεια των ενδιαφερομένων κλπ. Μπορούν μερικά πράγματα να βελτιωθούν, αλλά θα ήθελα να αρχίσω λίγνοντάς σας τι ήδη υπάρχει. Πρώτα διαφάνεια και μετά για την υποπτία. Λοιπόν, όπως ξέρετε, η δημοσιονομική εποπτεία της Κομισιόν βασίζεται στις δημοσιονομικές της προβλέψεις. Δημοσιεύει τακτικά αναχώρα αναλύσεις των οικονομικών προοπτικών. Εκτός αυτού, μία φορά το χρόνο γράφει εκθέσεις με συνοπτική περιγραφή της κατάστασης και αναλύσεις για μακροοικονομικές τυχόν ανισορροπίες καθώς και αναλύει τους κύριους τις κύριες προκλήσεις, ιδιαίτερα για τη δημοσιονομική εποπτεία. Οι αξιολογήσει της Επιτροπής βασίζονται σε τεχνικές αναλύσεις που προετοιμάζουν οι υπηρεσίες τις δημόσιες και αυτές. Και όλα τα αποτελέσματα δημοσιεύονται στο, στην ιστοσελίδα της. Όλα τα στοιχεία δηλαδή που χρησιμοποιούνται από εμά είναι δημόσια διαθέσιμα. Φυσικά μπορούμε να διευκολύνουμε την πρόσβαση σε αυτές τις πληροφορίες και σας ευχαριστώ που βάλατε το θέμα θα ήθελα δεν να σας ανακοινώσω με χαρά ότι θα υπάρξει και μία νέα μορφή αυτή τη στιγμή των κανόνων για, τις ανα... κανόνες, των αναπτυξιακών κανόνων, το οποίο γνωρίζουμε εμείς στη γλώσσα μας ως βαντεμέκουμ ώστε οι χώρες με υπερβολικά ελλείμματα να είναι βέβαιο ότι έχουν πάρει τα μέτρα που χρειάζονται. Αυτά είναι τα τεχνικά στοιχεία των αναλύσεων και θα, τα οποία κυρώνονται στη συνέχεια από το σύνολο του Κολεγίου των Επιτρόπων. Όλα αυτά και οι πλήρεις πληροφορίες μπορούν να βρεθούν στην ιστοσελίδα μας όπως σας είπα. Γνωρίζουμε όμως και την ανάγκη για μεγαλύτερη αποσαφήνιση και θα κάνουμε κάτι για να βελτιωθεί αυτό. Όταν εξετάζουμε τη διαδικασία λήψης αποφάσεων της Κομισιόν, φυσικά οι αποφάσεις είναι πολιτικές, αλλά βασίζονται σε ανεξάρτητες αναλύσεις των στοιχείων και των κανόνων. Επομένως η Επιτροπή δεν μπορεί να αλλάξει τον κανόνα του 3% ελλείμματος ούτε το σύμφωνο σταθερότητος γιατί αυτά είναι στις συνθήκες τον οποίον θεματοφύλαξη είναι η Κομισιόν για την ελαστικότητα έχουμε κάνει μία ανακοίνωση για να γνωρίζουν οι χρήστες καλύτερα ποιοι κανόνες ισχύουν αντί να αλλάξουμε τους κανόνες πράγματι επειδή είναι πολύπλοκες οι καταστάσεις που αναλύουμε οι ρήτρε του SGP αφήνουν μεγάλα περιθώρια ερμηνείας και προς εσάς και προς το Συμβούλιο για να υπάρχει προβλεψιμότητα. Γι' αυτό μέσα στην εντολή μας είναι και το να κάνουμε ερμηνείες τους χωρίς να αλλάζουμε ή ανακαθιστούμε τους κανόνες για την σωστή δημοσιονομική διαχείριση. Α, είναι απαραίτητοι οι κανόνε αυτοί για να υπάρξει η νομισματική ένωση και γενικότερα για βιώσιμη ανάποτηξη. Και ακόμα σημαντικότερη είναι τώρα που πρέπει να αποφύγουμε την επανάληψη λαθών του παρελθόντος τις οικονομικές μας αναλύσεις τις δημοσιεύουμε αναχώρα τρεις μήνες νωρίτερα από ό,τι στο παρελθόν. Επίσης έχουμε διάλογο με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο στα πλαίσια του διμέτρου και του εξαμέτρου. Και τα μαθαίνει αυτά και ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Κυρίε και κύριοι, συμπερασματικά, η Κομισιόν είναι δεσμευμένη να επιτηρεί τους κανό την εφαρμογή των κανόνων. Ευχαριστώ. Ε, ευχαριστώ πολύ κύριε Επίτροπε και τώρα ακολουθούν οι ομιλητές εξ ονόματος των πολιτικών ομάδων. Θα σας παρακαλούσα αγαπητοί συνάδελφοι και πάλι να κάνουμε ησυχία για να ακούμε τους ομιλητές. Και θέλω να σας ενημερώσω ότι δεν υπάρχουν γαλάζιες κάρτες φυσικά αυτή τη στιγμή, ούτε catch the eye. Ο κύριος Ρωσάτη έχει το λόγο. Thank you, Madam Chair. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Επίτροπε, το Σύμφωνο Σταθερότητας και Ανάπτυξη είναι σημαντικό εργαλείο για να εξασφαλίζεται δημοσιονομική πειθαρχία στα κράτη-μέλη. Ε, καθ' τη διάρκεια της συζήτησης απόψε όμως τι είδαμε. Ούτε τα μέλη του Κοινοβουλίου, ούτε τα κράτη-μέλη είναι ευτυχισμένα και ευχαριστημένα με την εφαρμογή του. Χαίρομαι πάρα πολύ που ακούω τον Επίτροπο Κατάινεν να μας υπόσχεται ότι θα βελτιωθεί η διαφάνεια και η αποτελεσματικότητα του Συμφώνου Σταθερότητας και Ανάπτυξης. Ένας τρόπος ή ένας δρόμος είναι ενδεχομένως να σκεφτούμε να προσθέσουμε στο βασικό μέτρο δημοσιονομικής πειθαρχία που είναι το έλλειμμα και κάποιες άλλες παραμέτρους όπως είναι ο λόγος του χρέους προς το ΕΕΠ. Το έλλειμμα είτε είναι γενικό, νομαστικό ή διαρθρωτικό ε, υποφέρει από σημαντικές αδυναμίες. Το έλλειμμα μας δείχνει μια εικόνα ε, περιορισμένη χρονικά, βραχυπρόθεσμη και δεν προβλέπεται η βιωσιμότητα μακροχρόνια της δημοσιονομικής πολιτικής. Άλλος λόγος, ε, το έλλειμμα εξαρτάται πάρα πολύ από κυκλικούς παράγοντες, από συγκυριακά μέτρα ad hoc και από διακριτικά μέτρα πολιτικής που παίρνουν μεμονωμένες κυβερνήσεις. Από την άλλη, το διαρθρωτικό έλλειμμα είναι μια μεταβλητή η οποία δεν μπορεί να παρακολουθηθεί άμεσα και εξαρτάται και από το ενδεχόμενο ε, ε, ε, παραγόμενο αποτέλεσμα που είναι δύσκολο να μετρηθεί και να παρουσιαστεί με έναν τρόπο πιστικό. Λοιπόν, ενδεχομένως μια δυνατότητα βελτίωσης της κατάστασης θα ήταν ε, να ε, έχουμε το λόγο χρέους προς το ΑΕΠ για να έχουμε πιο μακροχρόνια πρόβλεψη της βιωσιμότητας της δημοσιονομικής. Ευχαριστώ κύριε Ρωσάτη. Ο κύριος Λούκ έχει τώρα το λόγο. Ένα λεπτό. Κυρία Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, με λίγο από αυτά που ακούω από τους προλαλήσαντες, διότι φέρεστε λες και υπάρχουν αντικειμενικές μέθοδοι. Δεν είναι θετική επιστήμη η οικονομία. Δεν είναι όλα μετρήσιμα με αυτόν τον τρόπο. Εγώ τα λέω αυτά ε, γιατί ήμουν και καθηγητής ε, εθνικής οικονομίας. Υπάρχουν πολλές διαφορετικές παραδοχές που μπορεί κανείς να χρησιμοποιήσει για αναλύσεις, ε, αριθμοί με παραμέτρους, με ε, υπολογισμούς που δεν μπορεί να είναι απριορή ε, ε, σωστή ή λάθος. Θέλουμε μεγαλύτερη διαφάνεια αλλά να μην εκινούμε από μία λάθος παραδοχή. Η εφαρμογή του Συμφώνου Σταθερότητας και Ανάπτυξης θα είναι ιστοδυναικές αδιαφανής. Θα πρέπει να το αναγνωρίσουμε. Από την ίδια του τη φύση είναι αδιαφανής και θα πρέπει να έχουμε κανόνες εύκολους να επιστρέψουμε στα βασικά στοιχεία της συνθήκης του Μαστρίχτ που είναι η ρήτρα μη διάσωσης. Ευχαριστώ. Thank you. The uh, ο κύριος Μπρίωρα για ένα λεπτό. Μπριουάμα. Ναι κυρίες και κύριοι το Σύμφωνο Σταθερότητας και Ανάπτυξης είναι πραγματική αποτυχία και θα πρέπει να ονομαστεί σύμφωνο αποσταθεροποίησης διότι η σταθερότητα υπάρχει για να εφαρμόζονται οι πολιτικές λιτότητας που χειροτερεύουν τα πράγματα που υποτίθεται ότι καταπολεμούν και έτσι εμποδίζεται κάθε αναθέρμανση της οικονομικής δραστηριότητας. Γι' αυτόν τον λόγο οι συστάσεις για τη διαφάνεια στην εφαρμογή του Συμφώνου Σταθερότητας δεν χρησιμεύουν σε τίποτα. Το παράδειγμα της Ελλάδας μας το έδειξε. Το παράδειγμα αυτό από την αρχή βασιζόταν σε δύο λάθος θέσεις. Την πρώτη, η πρώτη ήταν ότι η αναθέρμανση βασίζεται αποκλειστικά σε πολιτικές λιτότητας και έπειτα η πεποίθηση ότι τέτοια προγράμματα θα μπορούσαν να εφαρμόζονται αδιακρίτως σε οποιοδήποτε από τα 28 κράτη-μέλη αντί να κλείνετε τα έθνη σε δημοσιονομικούς και νομισματικούς κανόνες που δεν εφαρμόζονται, καλύτερα θα ήταν να προσπαθήσετε να δώσετε μια νέα πνοή στις οικονομίες των χωρών μελών που έχουν πρόβλημα για να μπορέσουν να βγουν πράγματι από την κρίση. Η επιστροφή της ανάπτυξης στην Ευρώπη θα εξαρτηθεί κυρίως από ριζιοσπαστική αλλαγή της οικονομικής και νομισματικής πολιτικής. Ευχαριστούμε. Επόμενος ο κύριος Μαριάς. Κοφίν εφαρμόζει το Σύμφωνο Σταθερότητας και Ανάπτυξης με δύο μέτρα και δύο σταθμά. Όταν πρόκειται για τη Γερμανία και τη Γαλλία κάνει τα στραβά μάτια, δίνει συγχώρο χάρτη και ανέχεται τις παραβιάσεις των κανόνων. Όταν πρόκειται για μικρές χώρες όπως η Ελλάδα τότε το ΕΚΟΦΗΝ επιβάλλει σκληρά μέτρα λιτότητας και βίες δημοσιονομικής προσαρμογής που φτωχοποιούν τους λαούς. Η Ελλάδα επί πέντε χρόνια βρίσκεται κάτω από τον ασφοκτικό έλεγχο και την εποπτεία της Τρόικας που έχει μετατραπεί σε σκυλό του Eurogroup και του ECOFIN. Το Σύμφωνο Σταθερότητας και Ανάπτυξης είναι ένα αντιδημοκρατικό εργαλείο με το οποίο επιβάλλεται απόλυτος έλεγχος στη δημοκρατική λειτουργία των κρατών μελών. Για να απαλλαγεί η Ελλάδα από την ενισχυμένη δημοσιονομική εποπτεία πρέπει να εγγράψει στον κρατικό προϋπολογισμό της τις οφειλές της Γερμανίας προς την Ελλάδα, δηλαδή τις πολεμικές επανορθώσεις και το αναγκαστικό κατοχικό δάνειο απαιτήσει ληξιπρόθεσμε και έντοκε που ανέρχονται σε 162 δισεκατομμύρια ευρώ συν του Γιατί η Ελλάδα είναι ο δανειστή και η Γερμανία είναι ο φιλέτη. Ευχαριστώ. Thank you. The next Ευχαριστώ. Επόμενο ομιλητή για ένα λεπτό, ο κύριο Μπονάνο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Νομίζω ότι είμαι σε ένα αμπαράκι και όχι στην Ολομέλεια του Κοινοβουλίου. Θα ήθελα να πω ότι παρά αυτήν την, τον συνεχή θόρυβο, να πω προς τον κύριο Κατάινεν ότι αν δούλευε σε ιδιωτική επιχείρηση θα τον είχαν απολύσει και αυτόν και τον Γιούνκερ. Οι Ηνωμένε Πολιτείε έχουν αναπτύξει την οικονομία τους προσπαθώντας να μειώσουν τους κανόνες και να αυξήσουν την ανάπτυξη. Εμείς στην Ευρώπη κάνουμε το αντίθετο. Ο γιος μου 12 ετών καταλαβαίνει ότι πρέπει να κάνουμε αυτά που κάνουν οι Αμερικανοί και όχι αυτά που κάνουν οι Ευρωπαίοι. Και δεν είναι ούτε πολιτικός ούτε οικονομολόγος. Το μοναδικό σύμφωνο σταθερότητας που μπορεί να υπάρξει στην Ευρώπη είναι για τους παράνομους, τους ε, παράτυπους. Αν το κάνουμε, αν το αποδεχθούμε αυτό θα λύσουμε το πρόβλημα γιατί αλλιώς η Ευρώπη από μόνη της τι να λύσει, τίποτα δεν μπορεί να λύσει. Θα δώσω το λόγο στον κύριο Κατάινεν. Δύο λεπτά παρακαλώ. Σας ευχαριστώ για αυτή την πολύ, την πολύ ζωηρή συζήτηση και ενδιαφέρουσα. Ο τελευταίος ομιλητής είπε ότι δεν υπάρχει κανένας κανόνας στην οικονομία και άλλοι πιστεύουν ότι θα πρέπει να υπάρξουν περισσότεροι και ισχυρότεροι και αυστηρότεροι κανόνες. Μιλήσατε όλοι όμως για την διαφάνεια στην εφαρμογή του συμφώνου. Είναι πολύ σημαντικό το θέμα αυτό. Ίσως ε, οι κανόνες να μην ήσαν ιδιαίτερα διαφανείς όσο έπρεπε και έχουν τεθεί πάρα πολλά ε, ερωτηματικά γύρω από την ερμηνεία που έχει γίνει στους συγκεκριμένους κανόνες. Κάποιοι πιστεύουν ότι ήταν πολύ χαλαρή η ερμηνεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, κάποιοι άλλοι ότι ήμασταν ιδιαίτερος ε, στενοί, αυστηροί. Γι' αυτό λοιπόν θα πρέπει να είμαστε προσεκτικοί στα θέματα της διαφάνειας. Όλοι θα πρέπει να κατανοήσουν τι σημαίνει σεβασμός στους κανόνες. Αν υπάρχει έλλειψη διαφάνειας, τι να σου κάνουν οι κανόνες. Και τότε οι κανόνες βέβαια είναι αυτοί που υφίστανται την κριτική. Προσπαθούμε να συγκεντρώσουμε την προσοχή μας στην έκθεση των πέντε προέδρων έτσι ώστε να προωθήσουμε περαιτέρω την αποτελεσματικότητα της πολιτικής μας. Προσωπικά θα μπορούσα να πω ότι η εφαρμογή των κανόνων είναι αυτό το οποίο μετράει. Όπως είπα νωρίτερα, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στα πλαίσια του ε, Συμφώνου Σταθερότητας έχει επιλέξει ένα ευέλικτο τρόπο εφαρμογής. Μπορούμε όμως να πούμε ότι παρόλα αυτά έχουμε σεβαστεί τους κανόνες αυτούς. Ένα από τα θέματα στα οποία δεν έχουμε δώσει πάρα πολύ προσοχή στο παρελθόν είναι το διαφθρωτικό κομμάτι της οικονομίας μας. Το θέμα δεν είναι το χρέος και το έλλειμμα. Το θέμα είναι επίσης και η ενίσχυση των δομών της οικονομίας και γι' αυτό θα ήθελα να στρέψουμε την προσοχή μας περισσότερο στη διαφθρωτική πλευρά της οικονομίας μας. Όταν βλέπουμε ποιες χώρες έχουν προβλήματα βλέπουμε ότι τα προβλήματα αυτά είναι πολλές φορές διαφθρωτικά και όχι κυκλικά. Γι' αυτό λοιπόν θα πρέπει οι παρεμβάσεις μας να έχουν ένα συγκεκριμένο στόχο, όχι μόνο πλαισίωση των επιμέρους προβλημάτων, αλλά να δώσουμε μεγαλύτερη προσοχή στο διαφθρωτικό κομμάτι. Σας ευχαριστώ. Πρόεδρε, η συζήτηση που προηγήθηκε ήταν όπως είπα ζωηρή και ενδιαφέρουσα. Ε, θα πρέπει να μην επανέλθουμε στο θέμα αυτό, θα πρέπει να προχωρήσουμε ακόμα περισσότερο στα θέματα αυτά. Σας ευχαριστώ. Θα δώσω τώρα το λόγο στην Καλίνα Λουκασέβιτσα για δύο λεπτά. Μόνο δύο λεπτά παρακαλώ. Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, κυρίε και κύριοι συνάδελφοι, χαίρομαι ιδιαίτερω και ευχαριστώ για την συζήτηση, η οποία δείχνει πόσο σημαντικό είναι να μπορέσουμε να φτάσουμε σε ένα καλό επίπεδο σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση με σταθερότητα και ανάπτυξη αηφόρο για την απασχόληση στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ύστερα μακροχρόνια στασιμότητα η Ευρωπαϊκή Ένωση χρειάζεται ανάπτυξη. Αυτή μπορούμε να την εξασφαλίσουμε με ταυτόχρονη υλοποίηση και της δημοσιονομικής ε, υπευθυνότητας και των μεταρρυθμίσεων των διαρθρωτικών και της σταθερότητας. Δεν είναι δυνατόν να μην επιτρέψουμε να επιτύχει το Σύμφωνο Σταθερότητας και Ανάπτυξης και η έκθεση των πέντε πρόεδρων που σήμερα αναφέρθηκε δείχνει ότι η οικονομική βιωσιμότητα και η ανάπτυξη είναι πάρα πολύ σημαντική και για την ανάπτυξη της ε, εμπιστοσύνης θα έχει πολύ μεγάλη σημασία το Σύμφωνο Σταθερότητας και Ανάπτυξης. Πρέπει να περιοριστούν οι κίνδυνοι για τα κράτη-μέλη και αυτό απαιτεί καταρχάς σημαντική οικονομική σύγκληση, δεύτερον σημαντική ενοποίηση των χρηματοπιστωτικών ε, αγορών και τις χρηματοπιστικές διατάξεις πρέπει να τηρούνται. Αυτό που είναι επίσης σημαντικό, θέλω να υπογραμμίσω, εν τέλει και που απαιτείται απαραίτητα, είναι να ενισχυθεί η πολιτική νομιμοποίηση και υπευθυνότητα. Γι' αυτό χρειάζεται πολύ στενότερη συμμετοχή των κοινοβουλίων των, των Ευρωπαϊκών Κρατών Μελών, του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, των κοινωνικών εταίρων. Έχουμε πολλά να κάνουμε από κοινού. Κυρίες και κύριοι βουλευτές, ολοκληρώνοντας τη συζήτηση αυτή, τελευταία για τη Λετωνική Προεδρία στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, θέλω να εκφράσω τις θερμότατες ευχαριστίες μου για την πολύ καλή συνεργασία και για τις συνομιλίες που μπορέσαμε να αναπτύξουμε εδώ από κοινού για το μέλλον της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σας ευχαριστώ θερμά. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστούμε την Προεδρία για την πολύ καλή συζήτηση που είχαμε και